από τις ομάδες cftd ENL και από τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές τα εξή αιτήματα διορισμών. Ο κύριος Ντονανό στη θέση του κυρίου Σαπρόν ως μέλος της αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης ε, των χωρών ΑΚΕ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος ο κύριος Ζακέ σε και ε, στη Λίμπε ο κύριος Σόσνιρς στη θέση του κυρίου Κορβιν Μίκε ως μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την ε, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας ο κύριος Τανάκης στη θέση του κυρίου Σαπρότ ε, στην ε, θέση της Επιτροπής Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάρχουν αντιρρήσεις